συντονιστές να δεχθούν τις ε, προτάσεις του εισηγητή του κ. Ρίκεϊ που αφορούν σε προγράμματα προτεραιότητες και προκατακτικές δράσεις και επίσης ε, επιθυμούν τέσσερα να επισημάνουν. Είναι το πρόγραμμα προτεραιότητας που έχει στόχο να βελτιώσει την βελτίωση συστημάτων ημέρωση των επιβατών και να απλουστευτεί η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων αυτά μέχρι μέσα από ένα ενιαίο ε, πολυγλωσσικό interface. Το άλλο είναι πρόγραμμα που αφορά στην ε, ε, πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ πρόκειται για θέματα στον τομέα του τουρισμού και επίσης να συνεχιστούν οι δράσεις που αφορούν στον βιώσιμο τουρισμό και στον τουρισμό τον κοινωνικό που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της, του προϋπολογισμού. Όσον αφορά την επιτροπολογία οι συντονιστές ε, αποφάσισαν ότι σε σχέση με τα μέτρα ως προς τη διαδικασία OPS ε, εκεί συμφώνησαν με την πρόταση της Κομισιόν να ορίσει, της Επιτροπής με συγχωρείτε, να ορίσει τον κύριο Γιαζεμπόφσκι εισηγητής για το σύστημα που αφορά στο Sky Packet. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έγινε πριν ε, ενημερωθούμε για την ε, Προεδρία της ε, Γερμανίας. Εντάξει, αστιάκι ήταν αυτό που είπα, μην το πάρετε σε σοβαρά. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι, ο παλιός καλός συνάδελφος, θα είναι ο συγητής και εκλήθη στην επόμενη συνεδρίαση για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά σε αυτά τα μέτρα. Και χαιρόμαστε που θα συμβεί αυτό. Στα διάφορα οι συντονιστέ έλαβαν υπόψη τους τι επιστολές τι οποίε εγώ έστειλα εξ ονόματό τους και ημών στον Επίτροπο κύριο Κάλλας ε, σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεταφορών εστάλει στη διάσκεψη των Πρόεδρων για τις ε, προτεραιότητες των μεταφορών όσον αφορά στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Εστάλει επιστολή στον κύριο Ταγιάννη ε, για το ατύχημα που έγινε με τον ποδηλάτη και σε σχέση με το γεωργικό εξοπλισμό και στείλαμε και μία επιστολή, ε, απάντησε ο πρόεδρος ε, Μπούζεκ ε, σχετικά με το θέμα του ότι οι εκθέσεις για τις μεταφορές ε, πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα ε, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και όχι να μεταφέρονται το βράδυ στη νυχτερινή ολομέλεια. Αυτό είναι ένα ε, πρόβλημα διαρκής. Εδώ και 20 χρόνια η Επιτροπή Μεταφορών ε, διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι στο Στρασβούργο παίρνει αυτό το σλότ το νυχτερινό ενώ η Επιτροπή ας πούμε, Εξωτερικών Υποθέσεων παρουσιάζει εκθέσεις πάντα το πρωί και ίσως θα πρέπει και αυτοί να μεταφερθούν το βράδυ. Πάντως θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό σλότ ε, στην Ολομέλεια για να μπορούμε να παρουσιάζουμε τις εκθέσεις μας. Επίσης, οι συντονιστές συμφώνησαν ότι στην επόμενη συνάντηση θα συζητηθεί το ενδεχόμενο συμφωνίας για τις ημερομηνίες σχετικά με την ε, παρουσίαση τροπολογιών ε, στην στον κατάλογο ψηφοφοριών. Αυτό προέκυψε από τη χθενή συζήτηση όπου είδαμε ότι είχαμε δυσκολίε με την τελευταία έκθεση για τη Γεωργία. Έτσι λοιπόν ε, την επόμενη φορά θα αλλάξει η κατάσταση. Αυτά είχα να σα πω από την συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να ρωτήσετε σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αν όχι, τότε ε, ευχαριστώ και προχωράμε. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση της κυρίας Αγιάλα Σάντερ η οποία τελικά τα κατάφερε να περάσει μέσα από τροπικές καταιγίδε, από την Τέφρα, να φτάσει από την Κεντρική Αμερική σήμερα εδώ για να μας μιλήσει για τα δικαιώματα των επιβατών στις και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Και μετά από αυτήν την έκθεση ε, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία των εκθέσεων. Η κυρία Αγιάλα Σάντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την κατανόηση και την υπομονή που έδειξαν οι συνάδελφοι. Γιατί δεν φανταζόμασταν όταν πάμε σε ταξίδι με προσωπία ότι θα επανέλθει η φύση με την εκδίκηση της κάτι που συνέβη. Βέβαια αφήσαμε τον πληθυσμό της Γουατεμάλα και του Σαλβαντόρ σε μια πολύ δεινή κατάσταση και μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν με την ελληνική φυσικά και των Ευρωπαίων. Θα ήθελα εντάχει να σας παρουσιάσω την κατάσταση σε σχέση με την έκθεσή μου. Είχα μια σειρά επαφών, πολύ καρποφόρων κατά τη γνώμη μου, με το Συμβούλιο, παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσία των σκιωδών εισηγητών. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε σημαντικές εξέλιξεις. Μια στιγμή, συγγνώμη κυρία Γιάλα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να περιορίσουμε λίγο το θόρυβο στην αίθουσα. Συγγνώμη κυρία Γιάλα, συνεχίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν έχουμε εντυπωσιακές εξελίξεις ως προς τη βελτίωση τη υλοποίηση του στόχου αυτού του θέματο, που είναι να κατοχυρώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τα δικαιώματα των επιβατών στις ε, θαλάσσιες μεταφορές, είτε σε κανονικά δρομολόγια, είτε σε κρουαζιέρες, είτε σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι ο στόχος, ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πρότασης. Δηλαδή να διασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα των επιβατών με ιδιαίτερη προσοχή στους επιβάτες με προβλήματα κινητικότητας. Στις μέχρι στιγμής προσπάθειές μου, εγώ προσπάθησα να εξομοιώσω την κατάσταση αυτή με τα δικαιώματα των επιβατών των αερομεταφορών και των επιβατών με ειδικέ ανάγκε, καθώ και τα δικαιώματα των επιβατών στι σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Προσπάθησα να εναρμονίσω κάπω την κατοχήρωση αυτών των δικαιωμάτων και αυτό έθεσα και στο Συμβούλιο, στις συνομιλίες μας και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες μου. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες των συναδέλφων, θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Κάποιοι συνάδελφοι διαπίστωσα ότι επιμένουν σε ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Μία τροπολογία, για παράδειγμα, προτείνει διατήρηση της πρότασης του Συμβουλίου, δηλαδή αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογή οδηγία των σκαφών που μεταφέρουν λιγότερου από 36 επιβάτες. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς τους συναδέλφους, ώστε στο μέτρο του δυνατού να εμείνουμε στην αρχική πρόταση του Κοινοβουλίου της πρώτης ανάγνωσης, που ούτω ή είχε συγκεντρώσει 568 ψήφους στην Ολομέλεια, μια σχεδόν συντριπτική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό προτείναμε, να περιλαμβάνονται όλα τα πλοία μέχρι 12 επιβάτες. Θα, θα σας θερμοπαρακαλούσα, συνάδελφοι, να εμείνουμε σε αυτή τη θέση της πρώτης ανάγνωσης. Γιατί είπαμε να αποκλειστούν οι πλωτές μεταφορές ποτάμιες μεταφορές που αντιμετωπίζουν κρίση. Αυτό το δεχτήκαμε. Και με την αποδοχή της πρότασης του Συμβουλίου να αποκλειστούν όσοι κυκλοφορούν σε απόσταση μικρότερη των 500 ε, μιλιών, μιλιών συμφωνήσαμε, αλλά παρακάλεσα να παραμείνουμε στο πεδίο εφαρμογή ε, και να διατηρήσουμε το όριο των 12 επιβατών. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους επιβάτες και υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης μέχρι την Ολομέλεια. Εμένοντας την πρώτη ανάγνωση μέχρι στιγμής καταφέραμε να περιορίσουμε αυτό το θέμα των, του εισιτηρίου για παράδειγμα. Θα υπολογιστεί η αποζημίωση με τρόπο που θα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα του κλάδου. Επίσης, βελτιώσαμε την προστασία των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Καταφέραμε να περιορίσουμε τις προθεσμίες ε, για την απάντηση, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να εμείνουμε και στο αρχικό πεδίο εφαρμογή αυτό που το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξε στην πρώτη ανάγνωση. Μην ζητάτε να παραταθεί το όριο στου 36 επιβάτες, παρακαλώ. Τουλάχιστον σε αυτή την ψηφοφορία, στην Επιτροπή, να εγκρίνουμε το... τις τροπολογίες 12 και 65. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες των κυρίων Βλάστο και Ρικέ που θα διαλευκάνουν την κατάσταση και θα διευκρινίσουν την νομική κατάσταση. Κυρία Μπιλμπάου, σας ευχαριστώ θερμά που με τις τροπολογίες σας επαναφέρατε τη θέση της πρώτης ανάγνωσης προς υπόμνηση, αλλά δυστυχώς πολλές τροπολογίες δεν θα μπορέσω να τις ε, εγκρίνω, γιατί προσπαθούμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις, ήδη έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε, οπότε μερικές τροπολογίες κυρία Πιλμπάου θα σας ζητήσω να τις καταψηφίσουμε, ενώ άλλες θα τις υποστηρίξω. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι θερμά τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις τους και να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι να παραμείνουμε στο πεδίο εφαρμογής της πρώτης ανάγνωσης με το όριο των 12 επιβατών και να ψηφίσουμε υπέρ των τροπολογιών 12 και 65. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις διαπραγματεύσεις μέχρι την Ολομέλεια δεν θα καταλήξουμε σε άλλες συμφωνίες. Αλλά προς το παρόν είναι σημαντικό ως διαπραγματευτικό εργαλείο να κρατήσουμε αυτή τη διαπραγματευτική θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αγιάλα. Η κυρία Βόρτμαν Κόλεκ, μέρος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γιαλασάντα η οποία παρουσίασε ένα πολύ καλό απολογισμό της κατάστασης και μας εξήγησε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Πριν λοιπόν αναφερθώ στα μεμονωμένα σημεία, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω μια γενική φύσεως παρατήρηση. Το ΕΛΚ στηρίζει το αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ορίζονται για ορισμένες ε, περιπτώσεις τα δικαιώματα των επιβατών για όλα τα μέσα μεταφοράς. και για τα λεωφορεία, για το θέμα για το οποίο είναι ο κύριος Κάντσια αρμόδιος. Εμείς λοιπόν ε, στηρίζουμε αυτή τη θέση και ως εκ τούτου η θέση, η εισήγηση της κυρίας Σάντερ είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Νομίζω ήδη κατά την πρώτη ανάγνωση ε, εξετάσαμε σε βάθος ε, την εισήγηση και το όλο θέμα και θα ήθελα να πεσημάνω στην κυρία Σάντερ ότι εμείς από πλευράς του ΕΛΚ ευθύς εξ αρχής πιέσαμε να υπάρχει κάποια αναλογικότητα στην έκθεσή της. Τι ακριβώς εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει ευελιξία κυρίως για τα μικρά σκάφη, για τις μικρές επιχειρήσεις ε, οι οποίες αναλαμβάνουν τις μικρές διαδρομές που έχουν άμεση επαφή με τους ε, επιβάτες. Και αυτό ισχύει και για τα αποκαλούμενα ιστορικά σκάφη όπου είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν ε, ορισμένα περιοριστικά μέτρα. Είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτές οι διατάξεις για να διασφαλιστεί η ε, πρόσβαση στα σκάφη. Εμεί ε, ταχθήκαμε υπέρ αυτού και γνωρίζετε, κυρία Σάντο, ότι τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες εμείς συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, γιατί έχω την αίσθηση ότι και το Συμβούλιο συμφωνεί μαζί μα. Δηλαδή και το Συμβούλιο ε, επιζητεί μια κοινή λύση η οποία όμως παράλληλα επιτρέπει και την απαραίτητη ευελιξία την οποία χρειαζόμαστε και εμείς για να μπορέσουμε να εφαρμόσει την οδηγία αυτή και στα μικρά σκάφη σε όλα τα κράτη-μέλη και να το πράξουμε αυτό ή δυνατόν χωρίς προβλήματα. Αυτή λοιπόν η ευελιξία πρέπει οπωσδήποτε να κατοχυρωθεί μέσα σε ένα ε, συμβιβασμό. Ε, λυπάμαι που δεν συνέβη κάτι τέτοιο μέχρι τώρα και αυτό το λόγο συνεχίζουμε τις επαφές. Ω εκ τούτου κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι εμεί. Ε, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις της εισηγήτριας. Υπάρχει όμως ένα θέμα καθοριστικής σημασίας. Πρόκειται για το πεδίο εφαρμογής. Ε, η οδηγία αυτή θα ισχύει για σκάφη με επιβάτες από 12 ή από 36 και πάνω. Αυτό είναι καθοριστικό, γιατί αν δεν αποφασίσουμε από αυτού, δεν διασφαλίζεται και η απαραίτητη ευελιξία. Ω εκ τούτου, η δική μου πολιτική ομάδα θα καταψηφίσει την τροπολογία υπαριθμών 12, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την εισηγήτρια να διεκδικήσει την απαραίτητη ευελιξία, από κοινού βέβαια με το Συμβούλιο. Και τα λέω όλα αυτά γιατί στο Συμβούλιο υφίστανται οι ίδιες ανησυχίες. Για μας αυτό είναι ένα καθοριστική σημασία θέμα και ως εκ τούτου εγώ ελπίζω ότι η ε, τροπολογία υπαριθμών 12 θα καταψηφθεί στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε κυρία Βαρτμανκόλη. Κυρία Μπιλμπάου για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που πολύ σωστά συνόψησε η κυρία Γιάλα αλλά θα ήθελα να πω ότι συνεργαστήκαμε πολύ στενά και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολλές επαφές τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να φέρουμε κοντά τις θέσεις μας και να προασπίσουμε τη θέση της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα τμήμα των τροπολογιών αντικατοπτρίζει αυτές τις συμφωνίες με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Νομίζω ότι το πιο επίμαχο θέμα είναι αυτό των επιβατών. Τα επιχειρήματα που ακούσαμε, δηλαδή ελαστικότητα αφενός και ιστορικός χαρακτήρας των πλοίων, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, νομίζω ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα απαντήθηκαν από την κυρία Γιάλα, γιατί το όριο των 500 μιλίων για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας ούτως ή άλλως αποκλείει τα πλοία αυτά που μεταφέρουν έως 12 επιβάτες ή λιγότερους. Συμφωνώ με την κυρία Γιάλα ότι θα πρέπει να μείνουμε στο όριο των 12 επιβατών γιατί γνωρίζουμε και τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, αλλά και οι σκιώδεις ηγητές ιδιαίτερα, ότι στην τελική απόφαση δεν θα μείνουμε στο 12, αλλά ούτε το 36 θέλουμε να δεχτούμε. Γιατί αναλύσαμε την κατάσταση στο κλάδο, είδαμε την πραγματικότητα που επικρατεί στην κάθε χώρα, είδαμε τι αντίκτυπο θα έχει μια κοινοτική οδηγία που θα προβλέπει ένα όριο 18 ή 24 επιβατών, γιατί ακόμη και αυτά τα όρια συζητήθηκαν στις ε, συνομιλίες με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Οπότε η συζήτηση είναι ανοιχτή, η διαπραγμάτευση δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε αν εμείς ψηφίσουμε το όριο των 12 επιβατών, έχουμε ένα καλό διαπραγματευτικό εργαλείο. Και έχουμε και δύο λόγους στα άλλα επιχειρήματα που ε, ανέφερα μερικοί, καλύπτονται από άλλα σημεία, ιδιαίτερα τα 500 μίλια. Και τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιείται αυτό ως ε, διαπραγματευτικό εργαλείο με την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το θέμα της υγείας. Εμείς είμαστε κατά της συμπερίληψης του θέματος της υγείας. Για να αποφευθεί η πώληση εισιτηρίων σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ή δυσκολίες κινητικότητας ή περιορισμένη κινητικότητα. Δεν θέλουμε η υγεία να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για άρνηση εισιτηρίου. Η άρνηση της πώληση εισιτηρίου σε οποιονδήποτε θα πρέπει να στηρίζεται σε λόγους ασφάλειας και σε καμία περίπτωση σε λόγους υγείας. Γιατί η νομοθετική αυτή διάταξη στόχο έχει να προασπίσει τα δικαιώματα και των ατόμων με αναπηρίες. Άλλωστε έχουμε επίγνωση ότι μερικές φορές είναι δύσκολες οι προσαρμογές αυτές, όχι μόνο για τα πλοία και για τα ξενοδοχεία, για τα μέσα μεταφοράς. Ε, για πολλούς λόγους, αλλά μεταξύ άλλων επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τέτοια προβλήματα κινητικότητας. Εμείς όμως θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια σε αυτή την πραγματικότητα και τις ανάγκες αυτών των ατόμων να τις περιλάβουμε σε όλες μας τις προτάσεις. Επαναλαμβάνω, εργαστήκαμε σκληρά, συμφωνήσαμε για πολλές τροπολογίες όπως φαίνεται και από τον κατάλογο. Ουσιαστικά επανήλθαμε σε μεγάλο βαθμό στην πρώτη ανάγνωση και η συμφωνία είναι αρκετά σημαντική. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι έγιναν διάφορες αλλαγές εκεί πέρα στην Επιτροπή. Άλλαξε η Γενική Διεύθυνση. Ο κύριος Κράμερ, 22 είναι σημαντική. Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά αυτή την επιχειρηματολογική αυτά που είπατε για τα άτομα με αναπηρία. Αποφασίσαμε για τα δικαιώματα ε, των επιβατών ε, στα πούλμαν, στα λεωφορεία και στις αεροπορικές στηρίες. Και είπαμε ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση αυτό το πληρώνουν όλοι οι άλλοι επιβάτες, ε, οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό να διατηρηθεί ως απόφαση. Και σας ανέφερα το παράδειγμα από τις ΗΠΑ Πολιτείες, όπου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ ήταν υποχρεωτικό σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ τα λεωφορεία να μπορούν να δέχονται απεριόριστα άτομα με αναπηρία. Αυτό δεν ήταν ε, λόγω συμπόνιας, αλλά λόγω των αναπήρων πολέμου. Για φανταστείτε λοιπόν, αυτό ε, πράγματι εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ. Ε, αν μπορεί να γίνεται στις ΗΠΑ, γιατί δεν μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί στην Ευρώπη. Και θέλω να μιλήσω και για τα ιστορικά οχήματα. Ε, τα ιστορικά οχήματα, αυτό είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι ένα πολιτιστικό αγαθό και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη τότε με τα ε, οχήματα αυτά. Πώς ε, οι άνθρωποι αυτοί πιέστηκαν γιατί δεν είχαν πρόσβαση. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι παράδειγμα έτσι ώστε το ίδιο να το εφαρμόσουμε και στα σκάφη. Να το εφαρμόσουμε σε αυτό το τομέα. Έχουμε λοιπόν την ε, τεχνολογία, την διαθέτουμε και στην περίπτωση αυτή ο επιβάτης είναι εκείνος που παίζει ρόλο και όχι το επιχειρηματικό κέρδος. Εάν λοιπόν επιβάλλουμε κάτι τέτοιο η κατάσταση θα αλλάξει άρδιν. Δεν μπορούμε κάθε φορά να ε, φέρνουμε σε μειονεκτική θέση τις, ε, τους σιδηρόδρομους και τώρα και τα σκάφη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι υπέρ ε, της ε, τροπολογίας και δεν θέλω η τροπολογία αυτή να απορριφθεί. Ο κύριος Έπη από τους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς, όχι, ο κύριος Κούν. Äh, Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στη συζήτησή μας. Εδώ ε, πρόκειται ε, για σκάφη και για τον αριθμό των επιβατών αν θα είναι 12 ή 36 όποιος λοιπόν ζει στην, ε, σε, ένα, σε μια παράκτια περιοχή και γνωρίζει το θέμα της ναυσιπλοείας γνωρίζει πολύ καλά ότι ε, υπάρχουν ε, και αυτές οι μερίσιες μετακινήσεις που προβλέπονται για όλους τους επιβάτες. Στην περίπτωση αυτή όπου δεν είναι η μετάβαση για τουριστικούς λόγους, αλλά για λόγους ε, καθημερινούς εξυπηρέτησης, τα εισιτήρια, τα αγοράζει κανείς επί τόπου και δεν τα έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως γνωρίζετε, θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα καταργήσουν διαδρομές. Αν... Ε, δεν είναι απολύτως σίγουρες ότι πράγματι οι επιβάτες διατρέχουν κίνδυνο. Σίγουρα τα ιστορικά σκάφη παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι το μέγεθος του σκάφους και η διαδρομή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι το Συμβούλιο και στη λυκή ανάλυση οι Υπουργοί Μεταφορών που θα ασχοληθούν με τα θέμα, αυτοί δεν το είπανε τυχαία αυτόν τον αριθμό των 36 επιβατών. Δεν πρέπει συλλήβδη να τα απορρίψουμε όλα, γιατί στην περίπτωση αυτή εμείς οι ευρωβουλευτές θα περάσουμε το μήνυμα προς τα έξω ότι προσπαθούμε να ε, επιφέρουμε μία ισοπαίδωση σε οτιδήποτε αφορά σκάφη που μεταφέρουν επιβάτες άνω τον αριθμό, πάνω από τον αριθμό των 12. Ε, υπάρχει το θέμα της αποζημίωσης, ε, της μη πρόσβασης Αυτά ε, θα πρέπει να διατηρηθούν, όπως ε, προβλέπετε βεβαίως ε, και στην αεροπλοεία και στους θεροδρόμους, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη. Και, εσύ, κύριε, και εσείς κύριε Κράμερ, φαντάζομαι θα γνωρίζετε ότι τα μικρά αυτά σκάφη που μεταφέρουν επιβάτες στον ποταμό Σπρέ ή κάπου αλλού, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, δεν μπορεί κανείς να τους επιβάλλει όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Ρεαλιστές πρέπει να είμαστε. Και αυτό σημαίνει πολιτική. Πολιτική σημαίνει να λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Ε, γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ όλοι εδώ ευρωβουλευτές να τα λάβουν αυτά υπόψη τους και να πάτε στις ε, πατρίδες σας ε, και να σκεφτείτε τι θα πείτε στους επιβάτες, τι θα πείτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Α, εσύ να πληρώσεις αποζημίωση σε αυτόν τον επιβάτη που δεν μπόρεσε να ανέβει σε ένα σκάφος γιατί φύσαγε φοβερός αέρας. Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος πως θα καταστραφεί η μικρομεσαία επιχείρηση αν του επιβάλλουμε τέτοιου είδου επιβαρύνσεις. Παρακαλώ πολύ να το σκεφτείτε αυτό. Ο κύριο Βαντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι υπέρ της ε, αναβάθμισης των δικαιωμάτων των επιβατών, ιδιαίτερα των επιβατών με περιορισμένη κινητικότητα Ευτυχώς κύριε Κράμερ δεν έχουμε παλέμαχος από το Βιετνάμ οπότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υιοθετήσουμε παρόμοιες διατάξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για το δεύτερο τμήμα το ιστορικό επιχείρημα δεν το κατάλαβα. Έχουμε εκατοντάδες, θα έχουμε εκατοντάδες, για ε, να μην πω χιλιάδες ε, ανέργους αν υιοθετήσουμε ένα τέτοιο μέτρο γιατί θα πολλαπλασιαστούν οι επιθεωρήσεις ε, στα πλοία αυτά και ορισμένα μικρά πλοία δεν αντέχουν ε, το οικονομικό βάρος αυτών των προσαρμογών. Αν εγκρίνουμε μια τέτοια διάταξη θα οδηγήσουμε στην χρεοκοπία εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε οικονομική κρίση, θα επιτείνουμε την ανεργία με ένα τέτοιο μέτρο. Εγώ είμαι υπέρ της τροπολογίας 64 της κυρίας Βόρτμαν Κόλ και άλλων. Ευχαριστούμε κύριε Βαντάλεν. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γέγκλε, να πω ως πρόεδρος μερικά πράγματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ την κυρία Γιάλα Σέντερ γιατί κρατάει αυτό το πάθος της ε, για τις μεταφορές. Σας ευχαριστούμε. Ξεπερνάτε ακόμα και το Μάικλ. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των επιβατών, ιδιαίτερα των επιβατών με αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα και της ανάγκης οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης. Γιατί μια νομοθετική ρύθμιση έχει αξία μόνο εφόσον είναι εφικτή στην πράξη. Είμαι κάπως σε δίλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αδιαφορούμε για τους επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα ή επειδή θα έχει πρόβλημα το πλοίο να κάνει τις προσαρμογές ή επειδή ένα πλοίο έχει ιστορικό χαρακτήρα. Έχει δίκιο ο κύριος Κράμερ, αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κούν. Θα πρέπει ε, να δούμε αν η ρύθμιση που προτείνουμε είναι εφικτή. Αν ε, επίσης μπορεί να την αντέξει οικονομικά ο επιχειρηματίας. Αναφέρθηκε το επιχείρημα των ιστορικών σκαφών. Όπως ξέρετε, ε, η δική μας ε, πολιτιστική κληρονομιά στις μεταφορές που είναι η σιδηρόδρομη, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοια μέτρα ε, για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Και μάλιστα η συμπερίληψη τέτοιων ε, μέτρων ενισχύει την κινητικότητα με τους σιδηροδρόμους και το ιστορικό επιχείρημα δεν ισχύει. Δεν ισχύει στους σιδηρόδρομους τουλάχιστον. Ο κόσμος επισκέπτεται περισσότερο όταν υπάρχουν, υπάρχει δυνατότητα με τις προσαρμογές αυτές να επισκεφτούν περισσότεροι άνθρωποι. Το ίδιο ισχύει και για το ιστορικό πλοίο. Δεν νομίζω ότι ο ιστορικός χαρακτήρας είναι επιχείρημα κατά των προσαρμογών αυτών για τους ε, ανάπηρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Πρόεδρο για την πολύ ισοσκελισμένη προσέγγιση που έχει, ζήτημα το οποίο το εκτιμά ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και όλους τους βουλευτές από την Επιτροπή Μεταφορών για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει προκειμένου να προασπίζονται περισσότερο τα δικαιώματα των επιβατών θαλασσίων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και την εισηγήτρια και βλέπουμε επίσης ποια είναι η στάση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμφωνία και θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δύο βασικά είναι τα ζητήματα εδώ πέρα όσον μας αφορά. Πρώτον, το πεδίο εφαρμογή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των συζητήσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικό τα δικαιώματα των επιβατών να καλύπτονται με όσο το δυνατό πιο ευρύ τρόπο. Γι' αυτό το λόγο προτείνουμε 12 επιβάτες ω όριο για το πεδίο εφαρμογή και γνωρίζετε βέβαια ότι η θέση του Συμβουλίου είναι 36 επιβάτες. Βέβαια, η σωστή λύση ενδεχομένω να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο αυτά όρια και περιμένουμε να δούμε και τη δική σα ψηφοφορία για να δούμε τελικά ποιο θα είναι αυτό το εύρο του πεδίου εφαρμογή που θα αποφασίσετε. Σα επαναλαμβάνω όμω και πάλι ότι το ζήτημα του πεδίου εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερου επιβάτε. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνουμε την έβρεση συμβιβασμού. Ε, το ζήτημα της υγείας είναι το δεύτερο σημαντικό ζήτημα, ιδίως όσον αφορά τα κρουαζιερόπλια. Θα πρέπει... Εδώ πέρα να καλύπτονται τα δικαιώματα των επιβατών εξίσου. Έχει ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η λύση πάλι θα πρέπει να βασίζεται στην μη διάκριση. Μια, ένα νέο άρθρο 4α υπάρχει εδώ πέρα, το οποίο θα πρέπει να ισχύει για όλους τους επιβάτες και να επιτρέπεται σε μεμονωμένες ε, υπηρεσίες να αρνούνται την επιβίβαση κάποιων επιβατών όταν ε, διακυβεύεται η ε, υγεία τους. Θεωρούμε ότι η λύση αυτή είναι καλή και νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα μια συμφωνία και από τις δύο πλευρές, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει τις επαφές της με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο προκειμένου να διευκολυνθεί η έβρεση συμφωνίας και με λίγη καλή θέληση, με λίγη καλή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση. Η λύση πιστεύω ότι βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογή τελικά και ζητάμε από τα μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών να καταφέρουν να καταλήξουμε το Συμβούλιο σε μια συμφωνία πριν από την ψηφορία στην Ολομέλεια. Πρόεδρος, ε, σας ε, ευχαριστούμε κυρία Γέγκλε που καταφέρατε να ε, βρείτε μία μέση λύση αν θέλετε να με στα δύο. Η κυρία Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να καθυσυχάσω όσους έχουν ακόμη φόβους ή επιφυλάξεις για την ελαστικότητα. Φοβούνται μήπως το κείμενό μου είναι άκαμπτο. Καταρχήν, οι ποτάμοι, οι συμπλωτές μεταφορές ε, αποκλείονται και προστατεύονται. Γιατί δεχόμαστε την πρόταση του Συμβουλίου για την ε, απόσταση των 500 μέτρων σε ένα δρομολόγιο. Επίσης, θα μπορούσα να δεχθώ ακόμη και την γερμανική τροπολογία να την υποστηρίξουν και άλλοι για να καθησυχάσω και τον κύριο Κούνε γιατί εκτός από τα 500 μέτρα που αποκλεί όλες ε, τις πλωτές μεταφορές για το Βερολίνο, το Πότσδαμ, όλες τις λίμνες σας διαβεβαιώ κύριε Κούν ότι αποκλείονται τέτοιες ε, πλωτές μεταφορές. Δεν είχα πρόβλημα με τη γερμανική τροπολογία. Τώρα, με το Συμβούλιο θα βρεθεί, ελπίζω, κάποια διάμεση λύση μεταξύ του ορίου των 12 και των 36. Να κρατήσουμε λίγο ευρύτερο το πεδίο εφαρμογή από το προτινόμενο από το Συμβούλιο. Αλλά ξέρετε πώ είναι οι διαπραγματεύσει. Αυτό είναι δεδομένο ότι αν ξεκινήσουμε από το 12 δεν θα σταματήσουμε στο 12. Κάπου ενδιάμεσα θα βρούμε τη λύση. Πάντως το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υπαναχωρήσει από την πρώτη στη δεύτερη ανάγνωση, γιατί στην πρώτη ανάγνωση που έγινε το 2009 υπήρχε συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του ορίου των 12 επιβατών. Ακόμη και το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι ήταν τότε υπέρ αυτού του ορίου. Και μάλιστα το Συμβούλιο ήταν ήδη πρόθυμο και ήδη είχε συγκεντρώσει πλειοψηφία για να εγκρίνει μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή και έκτοτε αναδιπλώθηκε και το Συμβούλιο εξαιτία αυτής της αλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα το Συμβούλιο χρησιμοποίησε αυτή την αλλαγή της θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δικαιολογήσει την πρόταση για τα 36. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, μην ξεχνάτε ε, ότι όλοι είμαστε ενδυνάμοι επιβάτε με περιορισμένη κινητικότητα. Δεν μιλούμε μόνο για του εγγενετεί ανάπηρου ή αυτού που είχαν κάποιο ατύχημα. Ο καθένα θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή να έχει πρόβλημα κινητικότητα. Γι' αυτό είναι λογικό να μπορεί ο κλάδο σταδιακά να προσαρμοστεί. Δεν υπάρχουν υποχρεώσει ούτε ριζοσπαστικέ ούτε δραστικέ. Αλλά να αρχίσουν σιγά σιγά τα πλοία ο ναυτιλιακός κλάδος ε, να προσαρμόζεται σταδιακά επαναλαμβάνω, βαθμιδών. Δεν πρόκειται για καμία ριζοσπαστική ε, υποχρέωση και διάταξη. Στο μέτρο του εφικτού φυσικά. Νομίζω ότι είναι και προς όφελος ε, του ναυτιλιακού κλάδου, γιατί ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γυράσκει, οπότε πολλοί άνθρωποι εξαιτία ηλικία του και τη περιορισμένη κινητικότητα, αν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλοία, θα σταματήσουν να ταξιδεύουν. Ούτω ή άλλω θα οδηγηθεί σε περιορισμένη απασχόληση ο ναυτιλιακό κλάδο, αν δεν κάνει αυτέ τι προσαρμογέ. Πιστεύω ότι αργότερα θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά να δεχτούμε από τώρα την πρόταση του Συμβουλίου νομίζω ότι θα μας ακινητοποιήσει διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ποτέ ανώδυνη μια πρόταση του Συμβουλίου. Άλλωστε, για όλα τα θέματα είπαμε να εμείνουμε στις προτάσεις μας. Και η περίφημη γερμανική τροπολογία ούτως ή άλλως είχαν προβλεφθεί για να εξασφαλίσουν αυτή την ελαστικότητα σας θέλω, παρακαλώ, ας εμείνουμε στην πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ακόμη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Και οι επιβάτες, αλλά και ο ίδιος ο κλάδος, γιατί είδαμε ότι και οι αερομεταφορές και οι σιδηρόδρομοι μεταμορφώθηκαν χάρη στι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όχι μόνο δεν υπήρξε απώλεια θέσεων απασχόληση, αλλά και βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες και έγιναν προς, πιο φιλικέ προ τον επιβάτη, έγιναν πιο ανθρώπινε, βελτιώθηκε η ποιότητά του. Γι' αυτό σα θέλω παρακαλώ, υπερψηφίστε τι τροπολογίε 12 και 65 για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο μέχρι την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάλα. Η ψηφοφορία θα γίνει τώρα. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω επίσημα και θα περάσει το θέμα στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, οι ψηφοφορίες. Θα αρχίσουμε με την έκθεση Καντσιάν. Αλλά πρώτα ας κάνουμε έναν έλεγχο της λειτουργίας των μηχανημάτων. Αν έχετε όλοι τις κάρτες σας παρακαλώ, ας κάνουμε τον έλεγχο. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. As everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, το ΕΛΚ έχει ε, μία παραπάνω ψήφων επιπλέον. So if you could sort that one out, Macho, as to who's not voting, because if Mrs. De Verac votes, then they've two. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί αν ψηφίσει τώρα και η κυρία Ντεβέρακ θα έχετε δύο επιπλέον ψήφους. Okay. Right, can we start? Πολύ ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το κατάλογο ψηφοφοριών. Ξεκινάμε τροπολογία 10 για την έκθεση Κάντσιαν. Άρθρο 2, παράγραφος 2, τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 του εισηγητή, όπου εδώ πέρα Ψηφίζουμε με την τροπολογία 1 on block για το σχετικό εκτιμώντας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 στη συνέχεια. Από τον εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν 62 και 63. Πάμε στην 14. Ξεχωριστή ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι το before by within three months υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, διαγραφή του 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, διαγραφή του και 6, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο είχαμε χωρίσει τη ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος. Όλοι ψήφισαν κατά τον ίδιο τρόπο και για τα τρία τμήματα. Άρθρο 2, τροπολογία 64 του κ. Μπράτμπουρν, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 του συγγήτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 καταπίπτει. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, η 65 δεν καταπίπτει υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66, 67, μαζί υπέρ, Είναι όλες οι ίδιες, λέει ο Πρόεδρος. Για ποιο λόγο έχουμε τρεις ταυτόσιμες. 66 με 70. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 71 74. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 75 του κυρίου Ούλμερ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 16, 17 και 2 μαζί οι τρεις αυτές τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 18 του συγητή ταυτόσημη με την 79 και μαζί με την τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 19, μαζί με τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 80, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21. Τροπολογία 21 είναι η επόμενη του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 καταπίπτει 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 85, πάμε στην 25 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 87 του κυρίου Φέρμπερ υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 88 του κύριου Μπράντμπουρν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 και 29 μαζί υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται. 90 της κυρίας Μάισνερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 του κυρίου Ούλμερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 92 καταπίπτει 32 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, διαγραφή του assistance to find. Δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε ψηφίζουμε για την 96 τροπολογία της κυρίας Σέρα Κιάνη άρχιτη ψηφοφορία αναφέρεται στο άρθρο 21 αυτή η τροπολογία έχετε τρεις επιπλέον ψήφους στο ΕΛΚ Το ECR, οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές έχουν μία επιπλέον ψήφο. Μπορεί το ΕΛΚΑ να βγάλει τρεις ψήφους, τρεις κάρτες και το ECR μία. Το ECR το έκανε, το ΕΛΚΑ βλέπω ότι είστε συν τρία ακόμα. Έχετε τρεις επιπλέον ψήφους. Μία επιπλέον έχετε τώρα. Νομίζω ότι ενδεχομένω ο συντονιστή θα πρέπει να θυσιάσει την ψήφο του. Μια χαρά είμαστε τώρα, ωραία. Πέρα ψηφοφορία. 24 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 33 καταπίπτει, πάμε στη 34. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 καταπίπτει, 98 της κυρίας Μάισνερ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 35 καταπίπτει. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101. ως επιπρόσθετη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 99 καταπίπτει. Πάμε στη 40 χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα διαγραφή του in accordance with national law και έπειτα το δεύτερο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 του συγητή υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 103 καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 40. Πάμε στην τροπολογία 38, λέει ο πρόεδρος, για το άρθρο 26, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 για το άρθρο 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 του κυρίου Φέρμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 του εισηγητή με προφορική τροπολογία που έχετε εδώ facilities on board υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο τροπολογία 49, εκτιμώντας 11, τροπολογία 49. Γιατί ήδη ψηφίσαμε την τροπολογία 1, μάλλον το σημείο 1 με την τροπολογία 11. Πάμε λοιπόν στην τροπολογία 49, Ντανέλης υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. η 50 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 52 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 52 σας παρακαλώ νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε για την τροπολογία 52 άρχιτη ψηφοφορία. Μη επιπλέον ψήφο έχει το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 6. Υπέρ. Υπέρ για την τροπολογία 6, λέει ο πρόεδρος κατά αποχές εγκρίνεται. Βλέπω ότι κουράζεστε σιγά σιγά και έχουμε πολλές ψηφοφορίες ακόμα. Καταπίπτει η επόμενη τροπολογία. Πάμε στην 7 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτη Πάμε στην 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ως προσθήκη τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Μία επιπλέον ψήφο έχει πάλι το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρας πληροφορίας. 36 υπέρ, ουδής κατά, 40 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κάνσιαν. Switch of modes. Change of operative. Αλλαγή φρουράς. Έρχεται ο καπετάνιος. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα δώσετε τις αρθρώσεις σας, άρθρο 2.1β, τροπολογία 63, Αγιάλα Σέντερ, έκθεση, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 και 65 πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 12 και 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος. 18 υπέρ, 16 κατά, 6 αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται οι τροπολογίες 12 και 65. Τροπολογία 64, Βόρτμαν Κόλ, ως προσθήκη. Ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ της 64. Κυρία Βόρτμαν Κόλ. Διαφωνώ ότι είναι προσθήκη. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ολόκληρο, ολόκληρη την τροπολογία. Γιατί και η 36 είναι μέσα. Είμαι κατά της α, ε, μόνο της τροπολογίας αυτής. Λάθος, ε, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Επειδή εγκρίθηκαν οι τροπολογίες 12 65, μόνος προσθήκη μπορεί να ψηφιστεί 64. Καλώς, καλώς, εντάξει. Έστω και ως προσθήκη. Ως προσθήκη, λοιπόν. Τροπολογία 64. Ποιος είναι υπέρ? Υπέρ της 64, Βαρτμαν Κόλ. Ως προσθήκη, επαναλαμβάνω, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 13 και 66 μαζί. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 13 και 66 άρχεται η ψηφοφορία PPE one too many again Thank you Mr Tartarelli and vote is closed ψηφοφορίας 21 ψήφισαν υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 15 και 67 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 68. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογίες 69 και 70 71, 72 και 73 Ευτόσιμες, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Άρθρο 3F, τροπολογία 74 της κυρίας Μπιλμπάου. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 76 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Το επόμενο βήμα είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο. Το βλέπω να έρχεται. 79. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. τέλο 21 υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται. 78, 80 και 81 καταπίπτουν. 82. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 82 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας 25 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Τροπολογία 83, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 86 άρχεται ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος 21 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 87 και 88 ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 91 άρχεται η ψηφοφορία The vote is open. I Τέλος. 13 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. 92. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 92. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 29 υπέρ, 11 κατά. Εγκρίνεται. 93. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα τροπολογία 98 Bradford Capping άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι τέλος 20 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται Τροπολογία 20 Ποιο Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 της ηγήτριας κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, το on request, κατά έτοιμο. Το δεύτερο, το υπόλοιπο. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Πρώτο τμήμα της 23, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 100 καταπίπτει. 24, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, 25 υπέρ, 24 εγκρίθηκε κατά, αποχές εγκρίνεται και 25. Αλλαγή συζήτησης, βαθιά αναπνοή, αλλαγή σελίδας, βαθιά αναπνοή, 101 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 101, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 21 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 102. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. «26. Ψηφίζουμε το if possible ως προσθήκη, αν είναι δυνατόν. Υπέρ κατά άποχες μάλλον απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε για καλό και για κακό ως προστίκη η τροπολογία 26 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας 20 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 27 της συγγήτριας για το άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο 1, α, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 103 ως προσθήκη με, την, με εξαίρεση των, των κρουαζιέρων τη στιγμή της α, ε, κράτης υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν πέντε της Μπιλμπάου υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 106 και 107 ταυτόσιμες. Μαζί λοιπόν ψηφίζουν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 106 και 7. Ποιος άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος. 23 υπέρ, 18 κατά. Εγκρίνεται. 108, ποιος είναι υπέρ. 108 επαναλαμβάνω, ποιος είναι υπέρ. Η 106 εγκρίθηκε. 23-18 από ό,τι θυμάμαι, λέει ο πρόεδρος, εγκρίθηκε. 108 Φλέκενστάιν, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι τέλος 26 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται τροπολογία 29 της ηγήτριας ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 ποιος είναι υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 34 καταπίπτει. 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 111 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα τα 90 λεπτά δεύτερο, λεπτά, ε, δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος 112 κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Η τροπολογία 37 καλύπτεται. 113. Βλάβει στο κερί και ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος. 22 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117 της κυρίας Βόρτμαν Κόλ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλος. 20 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 40, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42. Συσχετίζεται με την 7. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα και πάροχη τελευματικών σταθμών και στις συνηθισμένες γλώσσες. Πρώτο τμήμα το 119, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45, ποιος είναι η 46 καταπίπτει, ποιος είναι υπέρ της 47,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 121 υπέρ, κα, κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 6 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 58 της κυρίας Λίχτεμπέργκερ. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά... Φαίνεται ότι έχει κουραστεί τα χεράκια σας. Τέλος ψηφοφορίας 22 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 4 της συγκίτριας ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται Έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 Ψηφίζουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, αυτή η πληροφορία μέχρι την ticketing. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 κατά καταπίπτει, 62 κόσα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20, 10 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τροπολογία 10 τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά As everybody voted, the vote is... Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 24 ψήφισαν υπέρ, μία ψήφος κατά και 17 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γιάλα Σέντερ. Right, what's this? Mrs. is Mrs. Deverac's report next. Επόμενη έκθεση Deverac. pages is it, this one? Yeah. Uh, are some so, uh, and oral amendments in the right. A and B. We have some Λοιπόν, έχουμε κάποιες ε, συμβαστικές ε, προτάσεις. Ε, το όλο θέμα είναι λιγάκι πιο περίπλοκο. Αν έχετε καλοσύνη, να δείξετε λίγη υπομονή. Ξεκινάμε με τη συμβαστική πρόταση 1 στο άρθρο 1. Είστε έτοιμοι όλοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, υπέρ της 1, παρακαλώ σηκώστε το χέρι, κατά, αποχές, γκρίνεται. Πάμε στην επόμενη Μαρινέσκου, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 86, Τικάου, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 88, Μαρινέσκου, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 90 91 92 ε, ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εγκρίνουμε. Τώρα υπάρχει έλεγχος. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. 26 υπέρ, 15 ε, κατά. 93 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 95 του κυρίου Ντεγκράντες. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96, 97, 98 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 αποσύρθηκε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 με προφορική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Εκατόν ε, σε τμήματα ψηφίζουμε πρώτο τμήμα μέχρι εκεί που λέει administrative proceedings και το δεύτερο τμήμα είναι η τελευταία πρώτη τροπολογίας Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται υπέρ για το δεύτερο τμήμα κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε ξέρω ότι είναι δύσκολο ε, να ψηφίζει κανείς όλα αυτά αλλά τι να κάνουμε για το δεύτερο τμήμα της 103 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι έκλεισε η ψηφοφορία 20 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 104 κυρία Λίχτενμπεργκερ υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 105 καταπίπτη, 106 βαντάλεν υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 107 Μαρινέσκου υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η 19 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 συγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 συμβατεί με την τροπολογία 22 έτσι ψηφίζουμε ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 23 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 0 καταπίτη, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφανώς ο κύριο Μαρινέσκου υπερψήφισε την τροπολογία του, το είδαμε αυτό. Η 111 σε τμήματα, πρώτο τμήμα, ε, μέχρι εκεί που λέει ε, Coordinator of the Network, δεύτερο τμήμα, μέχρι εκεί που λέει Substantiated. Πρώτο τμήμα ε, της 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται η 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 30 αποσύρθηκε. 31. Εισηγητής. Άρθρο 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 115. κάω, Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 33 εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 κυρίως Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 36 εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 120 είναι η προσθήκη, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 124. 124 και 127 να τις πάρουμε ε, μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 129 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 130 ε, και την 131. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 130 και την 131. Ε, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Η 40 καταπίπτει, η 132 καταπίπτει. Πάμε τώρα στην 133. Σε τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι ε, to disclose και δεύτερο τμήμα which it is authorized to disclose μέχρι εκεί και θα καταπέσει έτσι και αλλιώ, καταπίπτει έτσι και αλλιώ, γιατί εγκρίναμε την 130, άρα ψηφίζουμε μόνο για το πρώτο τμήμα. Συμφωνείτε, το πρώτο τμήμα λοιπόν, 133, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 επίσης ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 41 ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 140 και 41 είναι πανομοιότυπες υπέρ κατά ε, αποχές ε, εγκρίνεται 44 λοιπόν καταπίπτει 142 ε, υπέρ κατά αποχές γκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην 143 και την 144 από κοινού ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά 143 και 44 από κοινού ως προσθήκη ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. 20 υπέρ. Απορρίπτεται και 145 ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Μισό λεπτό. Η 47 καταπίπτει. Ψηφίζουμε για την 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 47 καταπίπτει 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται από 48 μέχρι 52 όλες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 151 σε τμήματα σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα ε, EU Airlines, δεύτερο τμήμα Making it possible before takeoff και τρίτο τμήμα, ε, πρώτο, τμήμα λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά εγκρίνεται 153 Βαντάλεν. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 22 υπέρ ε, γκρίνεται. Τώρα η 55. Η 56 Πριν ψηφίσουμε την 56 θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η τροπολογία αυτή που ζητά έναν άτομο, ένα άτομο σημείο επαφής σε περίπτωση ατυχήματος υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Φορέα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτό απλώς θέλω να πω για να καθησυχάσω τους συναδέλφου από διάφορες πολιτικές ομάδες. Πολύ ωραία. Η 56 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 57 αποσύρθηκε, η 157 είναι η επόμενη υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Κυρία Αλβάρες, ε, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Πάμε στην 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 58. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 ε, από τον κύριο Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 το δεύτερο τμήμα γιατί το πρώτο τμήμα καταπίπτει λόγω της 160. Ε, ε, το δεύτερο λοιπόν ε, τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. «162 De Grande προσθήκη υπέρ παρακαλώ». «Κατά αποχές εγκρίνεται». Η 163 καταπίπτει. Η 60 του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. η 62, 63, 64 ενσώματοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 164 μέχρι την 167 ε, να ψηφίσουμε για όλες αυτές μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 170 του κυρίου Μαρινέσκου. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα του 69 έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε μόνο για το δεύτερο τμήμα της 69 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω απορρίπτεται, αλλά ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 69. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει. Ψηφίζουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 καταπίτη. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 72 καταπίπτει, 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει, η 74 καταπίπτει, 75 επόμενη υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε την 75 ψηφίζουμε. Ψήφισατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία 18 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. Η 5 εισηγητής κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 6 6,76 και 7 από κοινού η 78 καταπίπτει, η 77 ως προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές, ε, θα ελέγξουμε. Η 77 ως προσθήκη ε, ψηφίζουμε. Ψήφισατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. 21 υπέρ, εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα του 79 καταπίπτει, το δεύτερο τμήμα ως προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εκρίνεται 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η, η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 82 σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα ε, είναι μέχρι information και το υπόλοιπο είναι το δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ του πρώτου τμήματος κατά αποχές ε, εγκρίνεται πάμε στο δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος του δεύτερου τμήματος του 82 ψηφίζουμε ψηφίσατε όλοι Απορρίπτεται. 12. Ε, έχει καταπέσει 11. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 83. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 13 έχει καταπέσει. 84. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ε, συγχαρητήρια κυρία Ντεβέιρακ. Επίσης... Ε, Έχουμε και το νομοθετικό ψήφισμα. Κατόπιν τούτου ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Ψήφισατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Το ίδιο αποτέλεσμα. 31 υπέρ, κανείς κατά μία αποχή για το νομοθετικό ψήφισμα και πάλι ε, συγχαρητήρια κυρία Ντεβέιρακ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι έχουμε και άλλες ψηφοφορίες, πάντως στις 11.30 έχουμε τριμερή συζήτηση για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να δοθεί επίσημη εντολή στην Επιτροπή μας, προκειμένου να καταφέρουμε με τους σκιώδεις εισηγητές να διαπραγματευτούμε με την Προεδρία του Συμβουλίου βάσει των όσων εγκρίναμε και ψηφίσαμε σήμερα το πρωί. Και αν καταλήξουμε συμφωνία στις 22 Ιουνίου θα ξανάρθω εδώ πέρα για να κάνω απολογισμό των πορισμάτων της ε, διαπραγμάτευσης και για να εγκρίνουμε τα αποτελέσματα της τριμερής συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Ντεβέιρακ, προφανώ έχετε την εντολή της Επιτροπής μας, ψηφίσαμε άλλωστε. Μπορείτε λοιπόν εσείς με τους και ηγητέ, βάσει εντολή αυτή να πραγματευτείτε στον τριμερή διάλογο. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κύριου Γκρός. Να αλλάξει πάλι φρουρά εδώ πέρα. Είμαστε έτοιμοι πολύ ωραία. Τροπολογία 1 με 6 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 11. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 του κυρίου Βαντάλεν υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 64. Νομίζω ότι εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος, αλλά ψηφίζουμε και ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία για την 64. 18 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. 66 είναι η επόμενη τροπολογία υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά, αποχές, Ας ελέξουμε την 70 σας παρακαλώ. Τροπολογία 70, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Ε, η Άλντε έχει μία παραπάνω ψήφο. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 της κυρίας Λίχτενμπέργκερ υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97. Υπέρ κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 97. Σας παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία για την τροπολογία 97. Ψήφισαμε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. 98. Του κύριο Αλμπερτίνη, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε για τροπολογία 100 παρακαλώ τροπολογία φιντάντσα άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαμε όλοι πέρας 15 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται 102 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 Χένις Πλάσσερτ υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε για την 110 σας παρακαλώ. Ψηφίσαμε. Τέλος. 19 υπέρ, 21 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 130. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 17 υπέρ, 23 κατά, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, Ας ελέγξουμε για την 139 σας παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 με προφορική τροπολογία του κυρίου Ελ Καντράουι. Σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ελ Καντράουι θα παρουσίαζε κανονικά την ε, προφορική τροπολογία. Εγώ όμως θέλω να αντιταχθώ σε αυτήν, μήπως πρέπει να πάρει πρώτα κύριος Ελ Καντράουι το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητήσαμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Μας είπαν όμως ότι δεν ήταν δυνατό σε συμβαστική τροπολογία να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα πρέπει αυτό να έχει τη σύμφωνη γνώμη όλων των συναδέλφων. Γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε προφορική τροπολογία. Θα ήθελα λοιπόν, καθότι δεν διαπραγματεύτηκα δεσμευθήκατε μαζί μας για την προφορική αυτή να μην ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Συμφωνώ με την ερμηνεία αυτή. Είναι αδιάσπαστη η συμβαστική λύση, αλλά έχουμε και την προφορική τροπολογία που έχει γίνει δεκτή. Οπότε και η ψηφοφορία κατά τμήματα είναι σωστή λύση. Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη. Αν υπάρχει αντίθεση στην προφορική τροπολογία δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ίσως ε, το διαδικαστικό να το ρυθμίσουμε ως εξής, να πούμε ότι η προφορική ερώτηση και η ψηφοφορία σε αιτήματα κατά πόσο στην δέχονται και τα δύο. Και τα δύο σε ένα. Κοιτάξτε, ε, εάν ο κύριος Ελκαντραουή θελήσει να δεχθεί αυτό εν είδη προσθήκης και εγώ, γιατί όχι, το δέχομαι και εγώ, όμως ε, να το υποβάλει ως προσθήκη. Well, ε, ik, ik, ε, ik heb dit omdat... κοιτάξτε, εγώ υπέβαλα αυτή την πρόταση με τη διατύπωση που έχει τώρα, γιατί αυτή η διατύπωση εκφράζει καλύτερα τη θέση μας. Και δεν μπορώ να δεχθώ τον συνδυασμό και τον δύο. Ως εκ τούτου, εγώ αποσύρω την τροπολογία μου, αν θέλετε οπωσδήποτε βέβαια να την ψηφίσετε παρακαλώ, γιατί ξέρετε εμείς μπορούμε να δεχθούμε και τη συμβαστική πρόταση όπως την είχε διατυπώσει ο εισηγητής. γιατί ε, με τη συμβαστική πρόταση σε μεγάλο βαθμό λαμβάνονται υπόψη οι επιθυμίες μας. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για τη συμβαστική πρόταση. Ε, ε, ορισμένα μέλη της πολιτικής μας ομάδας δεν θα τη δεχτούν, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της αντίδρασης των φιλελευθέρων. Μάλιστα, λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση. Έχουμε μια συμβαστική τροπολογία αν έχουμε προφορική τροπολογία, τότε πρέπει να ξέρετε ότι η προφορική τροπολογία μπορεί να εισαχθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων της Επιτροπής. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Οι φιλεύθεροι λοιπόν είστε κατά αυτής προφορικής τροπολογίας. Αν ναι, τότε ψηφίσουμε απλώς τη συμβαστική 21 ως έχει. Αυτό κάνουμε υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται και στην Ολομέλεια βέβαια μπορεί να τροποποιηθεί εκ νέου, εφόσον αυτό αποφασίσουν οι συνάδελφοι. 141. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε συμφωνήσει για τη συμβαστική 21. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 150. Άρχεται η ψηφοφορία 150. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται ισοψηφία. 153 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική μάλλον 154 λέει ο πρόεδρος. 154 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 164. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας. 26 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 172 πέρας 15 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αποσύρεται 180, συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 183. Ξέρω ότι κουράζεστε σιγά σιγά με τις ψηφοφορίες, ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 183. Τέλος. 20 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 189. Ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε σας παρακαλώ για την 189 του κυρίου Ελκαντράου. Η άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 196 του κύριου Βαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε για την 197 σας παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία πρόκειται για τροπολογία του κύριου Βλασάκα Πέρας. 12 υπέρ 27 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 ράνερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 του κ. Βαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 245. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 246, ράνερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 247, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 249 ως παράγραφος 11α θα τοποθετηθεί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 254. Ξεχωριστή παράγραφος 14α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε για τη 254. Σας παρακαλώ. Ελεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 με 21. Η 256 το πρώτο τμήμα έχει καταπέσει. Πρέπει όμως να ψηφίσουμε για το δεύτερο τμήμα της 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ελέγχουμε τη 261. Άρθε ψηφοφορία για τη 261. Πέρας. Εγκρίνεται 20 υπέρ και 18 κατά. Πολύ καλά κάναμε που ελέγξαμε. 262 της κυρία Τικάου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 264 και 265 είναι πανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 267. Έχουμε εδώ προφορική τροπολογία από την κυρία Wortman Κολ Τη βλέπετε εδώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 267 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 268, ήταν ε, γλωσσική η τροπολογία που έγινε εδώ. Πάμε συμβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για τη 278. 278 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 15 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται. 279 του κύριου Βαντάλεν υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογή 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 33. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 295 ως προσθήκη υπέρ. Κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για τη 295. Τέλος. 17 υπέρ, 22 κατά, όντως απορρίπτεται, 299 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε για την 300. Αρχής ψηφοφορία. Τέλος. 19 υπέρ, 19 κατά απορρίπτεται. 303 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογή 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 311 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 315 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 327 Τροπολογία Γκρίσμπεκ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 332 της κυρίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 334 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 338 του κυρίου Ελ Καντράου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 339 λοιπόν. 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 344. Νομίζω ότι απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος, άρτη ψηφοφορία για την 344. Πέρας. 15 υπέρ, 25 κατά, όντως απορρίπτεται. 345 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 348 και 349 είναι πανομοιότυπες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 347 του κυρίου Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 355 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 359 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 369 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 371 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 372 και 373 είναι επανομοιότυπες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 1. Ένα λεπτάκι να τη βρω, λέει ο πρόεδρος. Σαν μαραθώνιος είναι αυτός που κάνουμε. Λοιπόν, συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 και 9 πανομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε για την τροπολογία 51 της κυρίας Γκουρμάη. Άρθιψη ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 20 κατά απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στις γνωμοδοτήσεις. Παράγραφος 4, γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μερικές βέβαια έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές λύσεις. NV4, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV7, παράγραφος 7. Δίκαια Δίκαιο μάθιο. Προσθήκη στην παραγράφα 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Εμβιεπτά MV7 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Παράγραφος 12. Συμφωνούμε ότι αυτή είναι η επόμενη ψηφοφορία για την παράγραφο 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα αναγοράζει το σύστημα εμπορίας εκπομπών, δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμβη 15. Δε, και νέα παραγράφος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 8 η επόμενη. Ποιος είναι υπέρ, Ήτρε παράγραφος 8. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Ήτρε 16 παράγραφος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αρχι... ε, της Περιφερειακής Επιτροπής 7, ΡΕΓΚΙ 7, πρώτο τμήμα για το μείγμα των μεταφορών, το βιώσιμο. Πρώτο τμήμα, Ρέγγι 7, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 7 Ρέτζι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι τέλος. 24 υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. Ρέτζι 9, δύο τμήματα και πάλι. Τονίζει τις ε, περιφέρειες με νησιά. Πρώτο, για τις περιοχές αρχιπελάγους, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δυστυχώς καταρρίφθηκαν οι περιφέρειες με αρχιπέλαγος. Απορρίφθηκε η τροπολογία. Δεύτερο τμήμα, ρεγγενέα, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα της ρέγγι 9. Ρέγγι 10, ψηφοφορία κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, χωρίς τις λέξεις και εντοπίζει αυτά τα αεροδρόμια. Δεύτερο τμήμα θα καταπέσει αν απορριφθεί το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ε, καλύτερα δεν μπορούσα να περιμένεις. Παμψηφί υπέρ, ούτε μία ψήφος κατά, ούτε μία αποχή. Συγχαρητήρια. Καλύτερο αποτέλεσμα ήταν αδύνατο. Μη φύγετε παρακαλώ γιατί έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Έκθεση Αλκαντράουι. Γνωμοδότηση μάλλον Αλκαντράουι. Change of personnel. Thanks for that, people. Αλλαγή φρουρά στο προσωπικό. Mr. Gross. Ο κύριος Γκρός. Κύριε Πρόεδρε, Ίσως είναι χρήσιμο ένα μικρό διάλειμμα. Είχαμε 400 τροπολογίες, ε, καταπληκτική συνεργασία, συλλογική προσπάθεια όλων των ομάδων. Σας ευχαριστώ θερμά όλους εσάς και τους συνεργάτες, τους βοηθούς και τη γραμματεία φυσικά, γιατί επαναλαμβάνω ήταν συλλογική προσπάθεια, πολύ δύσκολο το έργο, τιτάνιο και μέχρι τελευταία στιγμή ε, επεξεργαζόμασταν τις συμβαστικές λύσεις. Θερμά ευχαριστώ. Όντως, όντως. Αυτό ισχύει για όλες τις εκθέσεις που ψηφίσαμε σήμερα, γιατί όλες με τον τρόπο τους ήταν περίπλοκες. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη γνωμοδότηση του κυρίου Αλκαντράουι. Είστε έτοιμοι? Δύο μας έχουν μείνει ακόμη. Αλκαντράουι και Σίμψον. Έτσι δεν είναι. Η τελική ευθεία. Εδώ είναι που χάνονται, κερδίζονται τα μετάλλια του μαραθώνιου. Τελική ευθεία. Μία τελευταία προσπάθεια. Υπέρ του 10 κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 καταπίπτει. Τροπολογία 12. Τσικάου σε συνδυασμό με την τροπολογία 3. 12 σε συνδυασμό με την 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Καταπίπτει. 18. Τσικάου. Προφορική τροπολογία. Ως ξεχωριστό άρθρο 8α νέο. Προφορική τροπολογία του εισηγητού την έχετε πάρει. Υπάρχουν αντιρρήσεις όχι. Ποιος είναι υπέρ με την προφορική τροπολογία κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Καταπίπτει. 5. Ποιος είναι υπέρ της 5. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα του του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κατά καταπίπτει δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισετε όλοι. Τέλος. Προς 39 <laughs> υπέρ, χωρίς κατά, χωρίς αποχές, ε, πλησιάζει ο κύριος Αλκαντράουι το καταπληκτικό ρεκόρ του κύριου Γκρός. Περνάμε στην επόμενη έκθεση του Προέδρου για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Να σας υπενθυμίσω κάτι που είπαμε χθε στη συζήτηση. Δύο προφορικές τροπολογίες για τις παραγράφους 1 και 2, που ουσιαστικά προσθέτουν τη Βουλγαρία στο κατάλογο των χωρών, αλλάζοντας τον αριθμό από 21 σε 22. Ελπίζω να μην έχετε αντίρρηση διορθώνεται στις τροπολογίες, αλλά έπρεπε να το κάνω και επισήμω. Παράγραφος 1, προφορική τροπολογία, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, η τροπολογία του Προέδρου που προσθέτει τη Βουλγαρία, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, Μαρινέσκου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Αλχαντράουι. Υπέρ. 22 προς 21. Αλλάζει πάλι. Προφορική τροπολογία ισχύει και εδώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 με 22. Από 21 σε 22. Η 7 καταπίπτει. Παράγραφος 4. Προφορική τροπολογία του Προέδρου. Το ίδιο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 8 του κυρίου Μπαχ, Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 10 και 11 Ταυτόσιμες. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνονται. 12 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά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 επενδύσεων μέχρι το πολλέ περιπτώσει και το δεύτερο τμήμα παρατρύνει τα κράτη-μέλη μέχρι να διατηρήσουν επαρκώ. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Υπέρ του δεύτερου τμήματο, κατά, απόχέ. εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. 23 Τη κυρία Τσικάου. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 24. Ποιο είναι υπέρ, κατά, εποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Μάικλ Κράμερ. Εάν ψηφίσουμε για το 25, ε, δεν θεωρώ ότι καταπίπτει 26, γιατί η διαφάνεια ε, δεν ε, αναφέρεται σε αυτή την τροπολογία του κ. Κουνάρα, δεν καταπίπτει. Καλώς, σας φτάσουμε πρώτα στο σημείο αυτό, Μάικ. Πρώτα την 25 να μην προδικάσουμε τίποτα. 25. Ποιο είναι υπέρ. Κουν. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε τώρα ούτω ή άλλω μπορούμε να ψηφίσουμε την 26. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ίδιο αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε και 26 δυστυχώς Μάικλ. 27 του κυρίου Κούν. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 και 30 ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 31. Υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 29 και 30. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 19 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτονται. 31 του κυρίου Αλκαντράου, Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α, Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Ζήλε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 42 42. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 42. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 21 ψήφι υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 45, έτσι. Του κύριο Γκρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 47 της κυρίας Τσικάου άρχιτη ψηφοφορία ψήφισατε όλοι τέλος 18 υπέρ 22 κατά απορρίπτεται αιτιολογική σκέψη α 1 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται και τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 38 υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές εγκρίνεται και σας ευχαριστώ. Okay. Where are we now? Intelligent? Yeah, we can do the taxes. Mrs. Jensen is there, and the acting director, Monsieur Paquet, is also there. Mrs. Jensen, I'm just going to give them a... Κυρία Jensen. αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. 12 παρατέταρτο παρακαλώ να επανέλθετε στην αίθουσα ένα μικρό διάλειμμα και παρακαλώ ραντεβού σε 5 λεπτά. Λοιπόν, συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Η κυρία Γιάννησεν θα μιλήσει ε, για τα ITS. Ε, ξέρω ότι περιμένατε ε, κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών μαζί με εμά και σε ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε τα πέντε λεπτά διάλειμμα. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι θαυμάζω την πειθαρχία ε, με την οποία οργανώσατε τις ε, ψηφοφορίες, άρα προφανώς σας άξιζαν τα πέντε λεπτά διάλειμμα. Αυτό λοιπόν που θα σας παρουσιάσω είναι τα ευφυή συστήματα μεταφορών και η σχετική νομοθεσία. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι όλη αυτή η ιδέα το νομοθετικό σκέλος ε, έγινε καταρτίστηκε έτσι ώστε να υπάρχουν προδιαγραφές και εξειδικεύσεις στον τομέα των μεταφορών, των οδικών μεταφορών, έτσι ώστε να προαχθεί η χρήση αυτών των συστημάτων. Πρόκειψε λοιπόν μια συμφωνία με όσους εργάζονται στον τομέα αυτό ότι πράγματι κάτι πρέπει να γίνει γιατί η αγορά δεν μπορεί να ρυθμιστεί μόνη της ε, δεν μπορεί να προβεί σε μεγαλύτερη χρήση αυτών των ε, συστημάτων, τα οποία θα μπορούσαν βέβαια να μας ε, ωφελήσουν με περισσότερο αποτελεσματικές αλλά και πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάναμε στο Κοινοβούλιο όταν η Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο της, το οποίο αποτελείται από ένα πρόγραμμα δράσης με διάφορες ενέργειες και επίσης και προτάσεις ε, για νομοθετικές ρυθμίσεις. Κατά κάποιον ε, τρόπο περιχαρακώσαμε αυτές τις ε, προδιαγραφές και τα πρότυπα και είπαμε οι προδιαγραφές και τα πρότυπα πρέπει να συνδεθούν με το πρόγραμμα δράσης. Δεν θα προσφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να εκπονεί ε, προδιαγραφές για οτιδήποτε σε αυτόν τον τομέα. Μετά λοιπόν την ψηφοφορία της πρώτης ανάγνωσης πριν από τις ε, εκλογές επιβεβαιώσαμε την ψηφοφορία πρώτης ανάγνωσης και μετά τις εκλογές έλαβαν χώρα πολλές ε, διαπραγματεύσεις με τη Σουηδική Προεδρία η οποία πραγματικά έκανε μια καταπληκτική δουλειά, προσπάθησε να πείσει το Συμβούλιο ότι εδώ χρειαζόμαστε νομοθετικές ρυθμίσεις. Τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούσαν να υπάρχει κανός είδους νομοθετική ε, ρύθμιση ε, και ανησυχούσαν για το κόστος, το οποίο όμως τελικά είναι αρκετά περιορισμένο σε σχέση με άλλες ε, επενδύσεις ε, σε υποδομές σε αυτόν τον τομέα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Και αυτή η συμφωνία έχει άμεση σχέση και ε, συμβαδίζει με την κατεύθυνση που έχει ορίσει το Κοινοβούλιο για τέσσερις ε, τομείς. Εμείς ε, από πλευράς Κοινοβουλίου επιλέξαμε τέσσερις συγκεκριμένες δράσεις για την συγκέντρωση δεδομένων, για τις πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια, για την ασφάλεια και αυτές οι δράσεις τελικά αποδείχθηκαν έξι, κατ' ουσίαν όμως είναι οι ίδιες ε, προτάσεις όπως αυτές που παρουσίασε το Κοινοβούλιο. Ε, βεβαίως θα διερωτηθεί κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η διαφορά είναι η εφαρμογή. Δηλαδή το Συμβούλιο δεν επιθυμεί ε, άμεση εφαρμογή των προτύπων και προδιαγραφών που θα προέκυπταν από τη δουλειά της Επιτροπής και αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι σε 12 μήνες μετά την εκπόνηση προδιαγραφών ή προτύπων με τη διαδικασία της συναπόφασης θα έπρεπε να αποφασίσουμε σχετικά με την εφαρμογή. Βρήκαμε λοιπόν μία λύση σε αυτό το θέμα ε, της εφαρμογής. Ίσως όχι τη βέλτιστη λύση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία λύση οι ε, προδιαγραφές θα εφαρμοστούν και θέλω να πω ότι το τελευταίο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ε, η συνθήκη της Λισαβόνας και ξαφνικά δεν μιλάγαμε πια για επιτροπολογία αλλά για ε, πράξεις κατά εξουσιαδότηση. Αυτή αφορούσε την μεταφορά των 20 των ζώων και μετά την, ε, τα ITS. Αυτά ήταν τα πιλωτικά προγράμματα στα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν η κατεξουσιοδότηση πράξης. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε μέσα σε αυτή την διάσταση των θεσμών για το πώς θα ερμηνεύονται η κατεξουσιοδότηση πράξης. Και τώρα καταλήξαμε σε μια λύση που είναι πολύ ικανοποιητική και την οποία συστήνω σε αυτήν την Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Προτείνω να υπερψηφίσουμε και να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να φέρω ένα τελευταίο πράγμα που αφορά ιδιαίτερα τους πράσινους. Ε, θα θυμάστε ο κύριος Κουστάτσε που δεν είναι πια εδώ, ο κύριος Κουστάτσε από τους πράσινους επικεντρώθηκε στο ότι τα ευφύ συστήματα μεταφορών δεν είναι ευφύ και κατέθεσε μια τροπολογία η οποία εγκρίθηκε στην Ολομέλεια. Αυτή η τροπολογία πέρασε μάλιστα και από τις ε, νομικές και τις γλωσσικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν μπορείτε να πείτε στον κύριο Κουστάτσε ότι ε, η τροπολογία του έχει περάσει και τα ευρωπαϊκά ευφύ ε, συστήματα μεταφορών δεν είναι ευφύ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που είπατε. Και θα ήθελα να επαναλάβω και εγώ αυτά που είπα προηγουμένως προς την κυρία Γένσεν και προς τον Σκιώδη Σιγητή για τη θαυμάσια δουλειά που κάνατε και τον τρόπο που αντιμετωπίσατε το θέμα. Πράγματι προέκυψε αυτή η θεσμική αντιπαράθεση για τι ε, κατεξουσιοδότηση πράξης και νομίζω οι συνάδελφοί μας ε, στην Επιτροπή περιβάλλοντο, είναι εκείνοι που μίλησαν για τα διαβατήρια για τα οικόσιτα ζώα. Πάντως αναγνωρίζω τη δουλειά που κάνατε εσείς ως εισηγήτρια και οι σκιώδεις ε, συντονιστές για να φτάσουμε ε, σε αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι λοιπόν ως ε, πρόεδρος Επιτροπής σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Ο κύριος Κοχ από το ΕΛΚ. Κοιτάξτε, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω, απλά θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπε η κυρία Γένσεν και βεβαίως εγώ, εγώ εκ μέρους της πολιτικής μας ομάδας προτείνω ανεπιφύλακτα να υπερψηφίσουμε αυτά που προτείνει η κυρία Γένσεν. Η κυρία Τικάου. Εγώ ε, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Γένσεν γιατί η κυρία Γένσεν ε, εργάστηκε σκληρά και πολύ αποτελεσματικά και εγώ λοιπόν προτείνω την έγκριση των εγγράφων. Έτσι καλλιώς αυτό ήταν πάρα πολύ απλό για μας γιατί εμείς επιθυμούσαμε από την αρχή μια αυτόματη εφαρμογή, μια ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Βεβαίω ε, δεν ήταν δυνατόν να περάσουμε αυτόματα σε εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, αλλά έχουμε τώρα ένα πλαίσιο και αυτό είναι η ε, βέλτιστη συμβαστική πρόταση στην οποία μπορούσαμε να καταλήξουμε η Επιτροπή ε, Διαπραγματεύσεων ε, κατέθεσε μια πρόταση στο Συμβούλιο και αυτό ήταν καθοριστική σημασία. Συγχαρητήρια λοιπόν κυρία Γένσεν. Τώρα πλέον έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την ε, ανάπτυξη τέτοιων ευφυών συστημάτων στον τομέα των μεταφορών και βρισκόμαστε στην αρχή αλλά ενός πολύ ενδιαφέροντα δρόμου και στο μέλλον φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες ε, Πολλέ ε, τέτοιου είδου ενδιαφέρουσε ε, συζητήσεις. Η κυρία Λίχνμπεράγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό που είπατε για τον συνάδελφο Κούστετσερ και θα του τα μεταφέρω αυτά που είπατε. Εμείς είχαμε συμφωνήσει ότι η ευφυΐα είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με όντα και όχι με πράγματα. Και θέλω να επενθυμίσω το εξή. Υπάρχουν τώρα δύο μελέτες που έχουν αποδείξει ότι όταν υπάρχει τεράστια τεχνική ασφάλεια αυτομάτως ε, ε, μειώνεται η προσοχή και αυξάνονται οι πιθανότητες για ανθρώπινο λάθος. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε κατά νου αυτό. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε για ε, τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Το τι θα γίνει τώρα με αυτά τα θέματα νομίζω ότι αυτό για μας θα καταδείξει το μέλλον και οποιοδήποτε τώρα διαπραγματεύεται για τέτοιου είδους θέματα πρέπει να διαφυλάτει ως κόριο οφθαλμού τα δικαιώματα του ε, Κοινοβουλίου γιατί το Συμβούλιο επιθυμεί να μας αναχαιτήσει. Και ως εκ τούτου εγώ συμφωνώ μαζί σας με αυτά που είπατε όσον αφορά το περιεχόμενο πράγματι ε, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, και είμαι και εγώ ε, σύμφωνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτόματη εφαρμογή. Εκ μέρους της Επιτροπής ο κύριος Πακέη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γένσεν για την έκθεση σας αυτή. Ξέρετε ότι το σχέδιο δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη και θέλουμε να έχουμε και εμείς το νομικό αυτό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να περάσουμε στη νέα εποχή της εφαρμογής των νεφιών συστημάτων μεταφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Γένσεν καθώς επίσης και γέννη την Επιτροπή Μεταφορών για την σημαντική πρόοδο που χάρη σε εσά έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε. Σας ευχαριστούμε και εσά πολύ, λέει ο πρόεδρος, που ήρθε εδώ πέρα πιο νωρί και καταφέραμε να καλύψουμε το ζήτημα αυτό νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Πολύ ωραία. Υπάρχει τίποτα άλλο που θέλετε να προσθέσετε. Πρέπει να έχουμε μία προθεσμία για τις τροπολογίες, έτσι προβλέπει ο κανονισμός. Ελπίζω όμως να συμφωνούμε όλοι ατύπως τουλάχιστον ότι δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες και ότι στις 22 Ιουνίου θα ψηφίσουμε. Στις 3 Ιουνίου πάντως είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 22 Ιουνίου και θα πάμε στην Ολομέλεια τον Ιούλιο κάποιες τυπικές πληροφορίες λοιπόν αυτές που έπρεπε να σας δώσω. Ελπίζω πάντως ότι δεν θα έχουμε τροπολογίες και ότι συμφωνείτε κι εσείς με την προσέγγιση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πρωινή μας συνεδρίαση. Θα επιστρέψουμε